Καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας συνεδρία, συνάδελφοι. Της Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι μια κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας με την Επιτροπή ΚΟΝΤ, την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών και χαίρομαι όλος ιδιαιτέρως πριν ε, καλωσορίσω ε, τους ε, προσκεκλημένους μας να χαιρετήσω την κυρία Γκρέσλε από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Ε, σήμερα Αποστολή μας είναι να συζητήσουμε την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με την ε, επισκόπηση των επιδόσεων της διαχείρισης των υποθέσεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα ευθύ αμέσως να δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Θα έπρεπε να παραγγείλουμε σαμπάνια κανονικά, διότι η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού πάντοτε προσπάθησε και πολλά χρόνια κιόλα ε, για να γίνει ε, αυτός, αυτή η επισκόπηση. Και ε, θα λάβει το λόγο ο κ. Σκάδιφ τώρα για την παρουσίαση της επισκόπησης αυτής και τον παρακαλώ να λάβει αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα σας παρουσιάσω την ειδική μας έκθεση για την, για την επισκόπηση των επιδόσεων, τη διαχείριση των υποθέσεων. Μία ομάδα την ανέλαβε και λάβαμε υπόψη βεβαίως τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιλέξαμε αυτό ως ε, επίκεντρο. Γνωρίζετε ότι ο σκοπός του δικαστηρίου είναι να ελέγχει την τήρηση ε, της ενωσιακής νομοθεσίας και έχει το, αποτελείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, και το Γενικό Δικαστήριο. Θα χρησιμοποιήσω τον όρο ECA για το Εγκτικό Συνέδριο, το ε, ΔΕΕ, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Δικαστήριο και ε, Γενικό Δικαστήριο. Και όταν ε, λέω δικαστήρια θα αναφέρομαι και στα δύο. Έχει καταργηθεί το δικαστήριο το διοικητικό, οπότε δεν αναφέρεται στη σημερινή μας συνεδρίαση καθόλου. Έχει έναν προϋπολογισμό περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου 2.100 άτομα εργάζονται σε αυτό. 74 δικαστές ε, που θα γίνουν 84, όπως επίσης και 11 γενικούς εισαγγελείς. Για προφανείς λόγους οι άνθρωποι αυτοί ε, δεν μπορούν ε, να δέχονται πολιτικές πιέσεις και πρέπει να υπάρχει και λογοδοσία με τον τρόπο με τον, για τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί το προπολογισμό και το κάνει αυτό το δικαστήριο στον ιστότοπό του κάθε χρόνο ε, υπάρχει μία ε, διαβεβαίωση σε σχέση με τους λογαριασμούς ε, ε, για την ε, χρήση των πόρων. Θέλουμε όμως μια ευρύτερη λογοδοσία και να δούμε τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας του δικαστηρίου, πώς τα δικαστήρια διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό με τρόπο που σέβεται την ανεξαρτησία τους και ε, το ότι πρέπει να παραμείνουν εκτός πιέσεων, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία τους. Ο στόχος, τους ε, δεν, ε, ο μας δεν είναι μόνο τα πορίσματα, αλλά να ε, υπάρχει και λογοδοσία. Όπως γνωρίζετε, το ελεγκτικό συνέδριο ασχολείται και με κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θέλουμε ως ελεγκτικό συνέδριο να υποβάλουμε τις συστάσεις μας και για τους δύο αυτούς οργανισμούς. Εξετάσαμε κατά πόσο οι διαδικασίες ακολουθούνται σωστά και αν θα μπορούσε ο ρυθμός επίλυσης των υποθέσεων να είναι ταχύτερος. Εξετάσαμε λοιπόν ε, περίπου 28.280 υποθέσεις ε, κατά το 2014-2015. Είχαμε πάρα πολλές συνεντεύξεις ε, με ε, το προσωπικό, ε, με τους υπευθύνους. Ε, επιλέξαμε περίπου 30 υποθέσεις για να τις ελέγξουμε περισσότερο λεπτομερέστερα, να δούμε για ποιο λόγο μπορεί να καθυστέρησε η επίλυσή τους ή να επηρέασε τη διάρκεια της επίλυσής τους. Έχουμε ένα δείγμα, ε, θέλαμε όμως να δούμε τι ε, παράγοντες μπορούσαν να επηρεάσουν ε, την επίλυση των υποθέσεων και χρησιμοποιήσαμε και τους δικούς μας πόρους, ήρθαμε σε επαφή με τους δικαστές, τους κάναμε ρωτήσεις σε σχέση με τη λειτουργία του δικαστηρίου αλλά και με τη διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας, κάναμε πολλές ερωτήσεις για τη λειτουργία του, κάναμε πολλές ερωτήσεις που αφορούσαν ειδικότερα τις υποθέσεις 2014 και 2015 γιατί προφανώς μας ενδιαφέρουν ε, ε, οι ε, ολοκληρωμένες υποθέσεις που έχουν τελεσιδικήσει μας ενδιαφέρει επίσης η ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων όταν ήταν μερικές φορές απαραίτητο να μην μας δώσουν κάποιες πληροφορίες ε, οι ε, δικαστές. Θεωρούσαμε ότι είναι περίπλοκο το, περίπλοκη η διαδικασία χειρισμού των υποθέσεων. Συγγνώμη κύριε Κάρντιφ, λέει ο Πρόεδρος, μήπως θα μπορούσατε να μιλάτε λίγο πιο σιγά για να μπορούν να σας παρακολουθήσουν και οι διερμηνείς. Ναι, θα, θα το κάνω και ε, θα προσπαθήσω μάλιστα να βελτιώσω λίγο και την προφορά μου. Έχουμε λοιπόν ε, διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα περίπλοκο σύστημα διαχείρισης, το οποίο όμως δουλεύει καλά. Ε, έχει γίνει μια προσπάθεια καλύτερης αποδοτικότητας. Ε, η διαχείριση των υποθέσεων θα μπορούσε όμως να καταστεί ακόμη καλύτερη. Να σας δώσω κάποιες στατιστικές, κάποια στατιστικά στοιχεία. Την περίοδο 2009 και 2010 υπήρχαν περίπου 560 με 630 νέες υποθέσεις που κατατέθηκαν. 2015 με 2016 ήταν πάνω από 700 και το Γενικό Δικαστήριο το πρώτο αριθμητικό στοιχείο είναι περίπου 600 ε, και για το 2015 με 2016 περίπου 900. Οπότε έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας σε μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά τις ε, ε, υποθέσεις που έχουν ολοκληρωθεί, που έχουν κλείσει, για το Γενικό Δικαστήριο περίπου 620 με 700 ετησίως και για τη δεύτερη περίεργο 15 με 16 δηλαδή, περίπου 2.000, περίπου 1.000. Ε, είναι λοιπόν πολύ περισσότερες οι υποθέσεις από το 2009-2010. Ε, η συνολική διάρκεια κατά μέσο όρο έχει μειωθεί από περίπου 20 μήνες σε 15 μήνες ε, στο δικαστήριο και στο Γενικό Δικαστήριο από 26 σε 19 την ίδια χρονική περίοδο. Ε, βέβαια το μείγμα των υποθέσεων έχει αλλάξει. Δεν λέω ότι είναι επιστημονική η διαδικασία, αλλά ε, κάνουν πολύ περισσότερα τα δικαστήρια με τους σπόρους που έχουν στη διάθεσή τους. Ε, λιγότερο εντυπωσιακό, το Γενικό Δικαστήριο έχει μια καθυστέρηση στις υποθέσεις πηγαίνουν πέρα από το ενδεικτικό τους χρονοδιάγραμμά τους ε, και ε, αυτό σε ποσοστό 90% ε, περίπου. Ε, θεωρήσαμε ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος προσπαθεί να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Έχει λάβει λοιπόν ε, σημαντική, έχει αναλάβει σημαντική δράση και σε επίπεδο διαδικασίας και σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος. Ε, έχει, υπάρχουν κάποια ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα σε κομβικά σημεία του κύκλου ζωής των υποθέσεων και δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα ε, χρονοδιαγράμματα, κάτι το οποίο φυσικά έχει οδηγήσει σε αξιοσημείωτη πρόοδο. Όμως, όπως λέμε σε κάθε περίπτωση, ε, υπάρχουν πάντοτε περιθώρια βελτίωσης. Ε, η διαδικασία διαχείρισης των υποθέσεων δεν είναι προσαρμοσμένη σε ανάγκες κάθε ε, υπόθεσης. Ο μέσος χρόνος διάρκειας υπόθεσης είναι περίπου ίδιος για κάθε υπόθεση. υπόθεση. Δεν λαμβάνεται υπόψη, ας πούμε, το περίπλοκο μιας υπόθεσης, τι προσωπικό μπορεί να απασχολήσει. Επίσης, ε, το σύστημα ανάθεσης των υποθέσεων είναι αρκετά ε, βαρύ, δεδομένων όλων αυτών των παραγόντων. Ε, έχουν ένα σύστημα ανάθεσης των υποθέσεων ένας ε, ευρύτερος στόχος ε, είναι να υπάρξει μεγαλύτερη βελτίωση, να μειώνεται ο μέσος όρος ε, διαχείρισης των υποθέσεων. Δεν μπορεί να θεωρηθεί εύλογος παρόλα αυτά. Τουλάχιστον αυτό έχουμε κατανοήσει. Θέλει να έχει ένα πιο λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των υποθέσεων. Υπάρχουν όμως παράγοντες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές για να αξιολογηθεί το πόσο, περίπλοκο είναι, πόσο περίπλοκη είναι μια υπόθεση ή τι χρονοδιάγραμμα πρέπει να έχει. Αυτό βέβαια εξαρτάται ε, και από τους ίδιους τους δικαστές. Είδαμε επίσης και την υποδομή γύρω από τη διαχείριση των υποθέσεων. Τα συστήματα πληροφορικής είναι περίπλοκα και βασίζονται σε μια απαρχαιωμένη βάση δεδομένων. Ε, υπάρχουν μερικά καινούργια υποσυστήματα τα οποία προστέθηκαν συν το χρόνο, όμως δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα που να υποστηρίζει τη διαχείριση των υποθέσεων. Λοιπόν αυτή η κατάσταση, δηλαδή ένα απαρχαιωμένο σύστημα με νέα υποσυστήματα πιο σύγχρονα, δεν είναι ασυνήθιστη, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Ο μακροπρόθεσμος στόχος τους είναι να έχουν ένα καλύτερο σύστημα πληροφορικής. Εμείς φυσικά το προτείναμε και το υποστηρίξαμε ως ε, ε, πρόθεση. Τώρα οι διαδικασίες μετάφρασης ε, και αυτές εξετάστηκαν γιατί σε οποιαδήποτε γλώσσα μπορεί να κατατίθεται το δικόγραφο δεν ε, ε, υπάρχει γλω, γλώσσα λειτουργίας μόνο τα γαλλικά, οι διασκέψεις γίνονται όμως τα γαλλικά. Εντός του δικαστηρίου υπάρχουν κάποιες προτάσεις να γίνει μια σχέση, να γίνει μια εκτιμήση κόστους ωφέλους για να χρησιμοποιείται στο Γενικό Δικαστήριο και άλλη γλώσσα πέραν της γαλλικής γλώσσας. Εμείς δεν έχουμε άποψη προσωπικά ως ελεγκτικό συνέδριο για το πόσο θα βελτίωνε αυτό την κατάσταση, αλλά βέβαια περισσότερη ενημέρωση είναι πάντα καλύτερη από λιγότερη. Οπότε καλό θα ήταν να υπάρξει αυτή η αξιολόγηση για να δούμε κατά πόσο ε, υπάρχουν απαραίτητα, τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουμε να βασίσουμε μια τέτοια απόφαση. Αυτά από εμά. Ευχαρίστω να ακούσω ερωτήσει. Η κυρία Γκρέσλε, σας ευχαριστώ πολύ. Ας πούμε ότι αυτά που είπατε ως αφετηρία δίνουν πολλές υποσχέσεις. Θα ε, προτιμούσαμε το δικαστήριο να έχει πρόσβαση στα έγγραφα. Το έγγραφο άλλωστε, δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο εννοώ. Το, ε, είναι δημόσια έγγραφα αυτά. Εγώ είμαστε άλλωστε και συγκίτρια για όλη αυτή τη διαδικασία. Το ερώτημα είναι ποια έγγραφα, σε ποια έγγραφα θα ήθελε να έχει πρόσβαση το ελεγκτικό συνέδριο και προς το δικαστήριο. Γιατί δεν προσφέρθηκε πρόσβαση στο ελεγκτικό συνέδριο, ούτε καν σε έγγραφα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι υπάλληλοι. Οι στατιστικές, κύριε Κάρντιφ... τις οποίες ε, μας υποβάλλατε... και θέσατε στη διάθεσή μας, δίνουν μια συνολική ετήσια επισκόπηση. Δεν έχουμε καν στατιστικές σε βάση μηνός, μηνία βάση. Έχετε εξαιρέσει μάλιστα τις τελευταίες υποθέσεις. Άρα, η επισκόπηση σε βάση έτους ε, σημαίνει σημαντικά μειονεκτήματα. Κάποιο ο οποίο αναμένει την κρίση στην υπόθεσή του δεν τον διευκολύνει αυτό γιατί έχουν εξαιρεθεί οι ε, μακροβιότερες υποθέσεις. Ποιες στατιστικές θεωρείτε ότι πρέπει να έχουμε στη θέση μας για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα άλλωστε δεν κατανέμεται ισότιμα μέσα στο δικαστήριο. στη Γερμανία οι δικαστές αξιολογούνται και σύμφωνα με την απόδοσή τους. Ερώτηση λοιπόν προς το δικαστήριο τώρα. Ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Πώς αξιολογείται την αποδοτικότητα των δικαστών και των εισηγητών δικαστών. Δεν υπάρχει case management για την ώρα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποια αριθμητικά στοιχεία για κάθε φάση της διαδικασίας και εκεί πίσω από τα στοιχεία αυτά μπορούν να κρύβονται κάποιες ελληματικές αποδόσεις. Θα ήθελα να ακούσω από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τώρα σε ποια χρονικά διαστήματα μπορεί να γίνει μια αυστηρότερη αξιολόγηση δικαστών και τμήματων. Άλλη ερώτηση. Χρονολογικά ε, με ποιον τρόπο επεξεργάζονται τις υποθέσεις τους οι δικαστές και δεν μιλώ για ε, διαδικασίες επίγοντος, μιλώ για τις άλλες διαδικασίες που δεν έχουμε βρει καμία πληροφορία. Υπάρχουν στατιστικές του backlog των καθυστερουμένων υποθέσεων, ανατμήμα και αν όχι γιατί όχι. Έχουμε επιτύχει μια σημαντική μεταρρύθμιση με διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών. Και εν ώψη τώρα αυτού του διπλασιασμού αριθμού των δικαστών διερωτώ με τι κάνουν όλοι αυτοί οι δικαστές εάν δεν έχει αυξηθεί η απόδοση. Ποιε εξειδικεύσει υπάρχουν τώρα μέσα στο δικαστήριο το ίδιο και τι άλλο σχεδιάζεται προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν ερωτήθηκαν συστηματικά άλλωστε ούτε οι εισηγητές δικαστές που παίζουν σημαντικό ρόλο μέσα στο σύστημα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ερώτηση λοιπόν προ το ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί δεν ρωτήσατε συστηματικά του εισηγητέ δικαστέ. Και υπάρχουν και ορισμένε ενδιαφέρουσε διαπιστώσει που πρέπει να μα απασχολήσουν. Πρέπει να τις συζητήσουμε. Για παράδειγμα, παράγραφος 38 που λέει ότι η αποδοχή και επεξεργασία των εγγράφων από το γραφείο του δικαστή ευθύνεται για ένα 80 και πλέον των καθυστερήσεων. Έχουν δηλαδή λίγου πόρου τα γραφεία των δικαστών για το δικαστήριο υπάρχει μια ενδιαφέρουσα επισήμανση. Οι διακοπές των δικαστών. Λένε οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς ότι ένας από τους λόγους καθυστερήσεων είναι οι δικαστικές διακοπές. Γιατί δεν μειώνονται τότε οι δικαστικές διακοπές. Νομίζω ότι ε, υπάρχει επαρκής χώρος για βελτιώσεις. Και το ενδιαφέρον στο έγγραφο είναι ότι καταδεικνύονται οι δυνατότητες βελτιώσεως. Αλλά όχι στο βαθμό ευκρίνειας που θα θέλαμε. Όποιος παρακολουθεί το έργο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θεωρώ ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα αν εφαρμόσει την, το περιεχόμενο της επισκόπησης. Το πρόβλημα μου είναι ότι η κυρία Γκλέσλε έθεσε όλες τις ερωτήσεις που είχα κατά νου. Μια ακόμη ερώτηση όμως, ε, αν μπορούμε να τις ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις. Να ακούσουμε και τον κύριο Μερίνιο Πίντο. Συμφωνείτε να ακούσετε όλες τις ερωτήσεις και μετά να απαντήσετε. Νομίζω η κυρία Τζαμπάλοβα ήταν η πρώτη. Ευχαριστώ και τους δύο Προέδρου και τα μέλη των δύο δικαστηρίων και τους Συναδέλφου. Ευχαριστώ το Ελεκτικό Συνέδριο για την εκθεσή του και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις λεπτομερεί απαντήσεις. Σημειώνω με ικανοποίηση ότι τα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει κάνει σημαντικές, ε, έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες ε, για να βελτιώσει τη διεκπαιρέωση των υποθέσεων. Ε, έχει μειωθεί ο χρόνος που αφορά την εκδίκαση των υποθέσεων. Όμως, θα ήθελα εγώ να επικεντρωθώ στο θέμα της ε, αποδοτικότητας και των επιδόσεων. Ε, σε ό,τι αφορά τις δικαστικές αρχές θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να έχουμε ποιοτικές ε, αποφάσεις σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η αποτελεσματικότητα και η καλή επίδοση θα έπρεπε να ειδωθούν από μία άλλη σκοπιά. Ίσως ε, θα ήταν ε, μερικές φορές ε, καλύτερο να καθυστερούμε και να έχουμε καλύτερες και ακριβείς αποφάσεις παρά να βιαζόμαστε και να έχουμε χειρότερες ποιοτικές αποφάσεις. Εδώ όπως ε, συμφωνούν και τα δύο όργανα, είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να υλοποιηθεί η κάθε υπόθεση σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανά υπόθεση. Έτσι λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε προθεσμίες που θα ανταποκρίνονται σε κάθε υπόθεση ε, καθώς η πολυπλοκότητα των υποθέσεων είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και αφορά όλη την ε, διαδικασία. Η ερώτησή μου και στα δύο δικαστήρια είναι ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με την χρησιμοποίηση των ανθρώπινων πόρων ως ένα σημαντικός δείκτης αποτελεσματικότητας και Επίσης, ε, ο δεύτερος δείκτης αποτελεσματικότητας έχει να κάνει με την χρήση των ανθρώπινων πόρων, την ποιοτική τους χρήση. Ο κύριος Μαρίνιο Πίντο. Θέλω να θέσω δύο-τρεις ερωτήσεις, πολύ θεμελιώδεις, βασικές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, οι ερωτήσει είναι οι εξής ποιος ε, είναι ο αριθμός δικαστών ε, τον, του κάθε δικαστηρίου και ποιος είναι ο προϋπολογισμός που δαπανάται ετησίως για κάθε ένα από τα δικαστήρια αυτά, ποιος είναι ο αριθμός των δικών που εκδικάζονται σε κάθε ένα από αυτά τα δικαστήρια και ποιος ε, είναι ο αριθμός των δικών για τις οποίες υπάρχει ε, απόφαση και ποια είναι η αναλογία αριθμός δικών προς τον αριθμό των δικαστών, δηλαδή πόσες υποθέσεις αναλογούν σε κάθε δικαστή ετησίως και ποια είναι η αναλογία προϋπολογισμός δικαστή, δηλαδή πόσο κοστίζει ο κάθε δικαστής στους Ευρωπαίους φορολογουμένους και τέλος, ποια είναι η αναλογία προϋπολογισμός δίκη, πόσο κοστίζει η εκδίκωση μιας υπόθεσης σε κάθε ένα από τα δύο δικαστήρια. Αν μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος και θα σας ευγνωμονούσα. Ευχαριστώ, κύριος Ζιέφκα. Όχι. Κύριε Ντελβό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάντοτε εντυπωσιάζομαι πολύ όταν ακούω τις ερωτήσεις Είναι πολύ στοχευμένε οι ερωτήσει από την Επιτροπή προπολογισμού. Και σα ευχαριστώ που κάνετε αυτό το έργο, γιατί εγώ πάντα πάντοτε σκεφτόμουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα τη δικαιοσύνη, γιατί διαφέρουν οι υποθέσεις μεταξύ του και είναι πλοκό το ζήτημα. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, μιλάμε για μια δικαιοσύνη ποιοτική. Μπορούμε να αξιολογήσουμε, να μετρήσουμε την ποιότητα των δικαστηρίων ε, και να το δούμε αυτό σε σχέση με τη μείωση του αριθμού ε, των ε, εφέσεων. Είναι μία ερώτηση, μάλλον των προσφυγών ακύρωσης. Μια ερώτηση που θέτω για να δούμε αν μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα. Έχω και μία ερώτηση εμείς ε, δύσκολα συμφωνήσαμε για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και είχαμε την εξής απέτηση να υπάρχει ε, ουσιαστικά μεγαλύτερο σεβασμός ε, στην ε, ισότητα των δύο φύλων. Πόσες γυναίκες δικαστές υπάρχουν και ποια είναι η αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σας ευχαριστώ και των προτέρων για την απάντηση αυτή. Πρόεδρος. Κοιτάξτε, εγώ όταν βλέπω εδώ τις αντιπροσωπείες που έχουμε, μάλλον θα δίσταζα να μιλήσω για εις εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Μόνο άνδρες βλέπουμε, λέει η κυρία Ντελβό. Και πρέπει να δούμε τι συμβαίνει όχι μόνο στους δικαστές, αλλά και σε επίπεδο προσωπικού στην γραμματεία, στους εισηγητές. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Εμείς πάντων, να σκεφτούμε και τι συμβαίνει και στο Κοινοβούλιο. Κυρία Χαουτάλα, ευχαριστώ. Χαίρομαι που κυρία Ντελβό έθεσε αυτή την ερώτηση, γιατί είμαστε πάρα πολύ σοβαροί ε, σε σχέση με αυτή τη δήλωση που υιοθετήθηκε από τα τρία θεσμικά όργανα για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Και είναι πολύ μακριά το δικαστήριο στην επιταξή αυτού και το ίδιο ισχύει και για το ελεγκτικό συνέδριο, όπω γνωρίζω. Μόνο πέντε γυναίκε υπάρχουν στο ελεγκτικό συνέδριο, όπω ξέρω. Και μακάρι να κάνω λάθο. Βέβαια, ο αντίκτυπος της μεταρρύθμισης, στην οποία όλοι συμφωνήσαμε, στο Γενικό Δικαστήριο είναι κάτι πολύ σημαντικό για το μέλλον, για την αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση σε σχέση με τον αντίκτυπο του Brexit στις επιδόσεις ε, του δικαστηρίου. Έχετε κάποια σχέδια ε, για το πώς θα κινηθείτε μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο κύριος Λεμπρετών, θέλετε μια ερώτηση. Ζητώ συγγνώμη που έφτασα αργά. Είχα ενηλυμένες υποχρεώσεις, θα ήθελα να είμαι εδώ. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά ουσιαστικά τα προδικαστικά ερωτήματα που είναι πολύ σημαντικά για σας. Μπορείτε να προβλέψετε μείωση των προδικαστικών ερωτημάτων στο μέλλον, στο βαθμό που ήδη έχετε δώσει πολλές απαντήσεις. Μπορείτε να σκεφτείτε ότι οι εθνικές δικαιοδοσίες από τις σημερινές σας απαντήσεις θα μπορούσαν να, να συμπεράνουν ε, πώς θα επιλύσουν τις μελλοντικές διενέξεις. Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με το μέλλον της γαλλικής γλώσσας στο δικαστήριο. Πιστεύετε ότι είναι μια γλώσσα που έχει ακόμη μέλλον ή θα πρέπει ως Γάλλος να ανησυχήσω για το μέλλον της. Ευχαριστώ. Αυτές ε, ήταν όλες οι ερωτήσεις. Ε, ίσως ο κύριος Κάρντιφ θα ήθελε να αρχίσει ε, με τις απαντήσεις και μετά να δώσουμε το λόγο και στο δικαστήριο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερος για τα έγγραφα τα οποία θα θέλαμε να είχαμε δει, θα θέλαμε να είχαμε πρόσβαση, θα θέλαμε να είχαμε δει λίγο περισσότερα έγγραφα που αφορούν την εσωτερική διαδικασία. Αυτή στιγμή έχει ανατεθεί υπόθεση σε ένα δικαστή. Δηλαδή υπάρχει μία περίοδος ε, από τη γραμματεία μέχρι το δικαστή που ήταν ανοιχτή, αλλά αυτή τη στιγμή έχει ανατεθεί η υπόθεση στο δικαστή. Ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για μας, γιατί θεωρείται ότι έχει μπει σε διαδικασία διάσκεψης. Ε, βέβαια, ε, το κάθε, ο κάθε δικαστής έχει το δικό του σύστημα, έχει το δικό του γραφείο, ε, ο δικαστής, κυρίως άντρες είναι, ο κάθε δικαστής έχει διαφορετικό τρόπο ε, εργασίας και δεν μπορούμε να έχουμε μία απάντηση που να ισχύει για όλους. Όσον αφορά τις στατιστικές και κατά πόσο δίνουν την ετήσια εικόνα, τη γενική ετήσια εικόνα, ναι, θέλουμε να έχουμε περισσότερες και πιο προσαρμοσμένες πληροφορίες ε, κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει στην πρόοδο που θα θέλαμε και για τις μεμονωμένες υποθέσεις ως ελεγκτικό συνέδριο δεν ε, προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των δικαστών. Εμείς ε, δεν ε, κάνουμε εξατομικευμένη αξιολόγηση επιδόσεων. Μερικές φορές βέβαια το κάνουμε, κάνουμε κάποιες συστάσεις όταν κάτι δεν πάει καλά σε έναν οργανισμό. Αλλά για τα επόμενα, για τα επόμενα μας βήματα δεν θα γίνει άλλη αξιολόγηση ε, του ε, δικαστηρίου. Είναι, ε, δεν υπάρχει στο πρόγραμμά μας. Έχουμε πάντως ένα σύστημα παρακολούθησης και κατά την παρακολούθηση θα προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσο οι συστάσεις που κάναμε για ένα βελτιωμένο, πιο στοχοθετημένο σύστημα, ένα καλύτερο σύστημα πληροφορικής που κρατά ένα ε, ιστορικό ε, και καταγράφει καλύτερα την εξέλιξη των υποθέσεων ε, θα μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο έχουν ακολουθηθεί αυτές οι συστάσεις. Τώρα το πώς λειτουργεί ο κάθε δικαστής διαφοροποιείται από τον έναν δικαστή στον άλλο τα ε, συστήματα εργασίας είναι παρόμοια. Ε, βέβαια ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση, γιατί έχει το δικό του γραφείο. Εμείς όμως βλέπουμε απλώς τη διαχείριση της υπόθεσης, ε, το κατά πόσο δηλαδή προχωρούν οι υποθέσεις, όχι κατά πόσο είναι σωστή η απόφαση. Όσον αφορά τώρα τον ρόλο του, των εισηγητών όλοι οι δικαστές, τα τμήματα των δικαστών είναι υπεύθυνοι ε, για κάποιες ε, υποθέσεις, ε, τη βαριά δουλειά την κάνουν οι εισηγητές όμως κατά την προετοιμασία των υποθέσεων, οι οποίοι επιλέγονται ξεχωριστά από, τους, από τον κάθε δικαστή και είδαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι λαμπρότατη νομική, ε, των οποίων η δουλειά είναι πάρα πολύ σημαντική για την ευρύτερη διαχείριση των υποθέσεων και του συστήματο. Σε μερικέ περιπτώσει είδαμε ότι υπήρχαν καθυστερήσει ε, γιατί δεν υπήρχαν ε, νομικοί διαθέσιμοι και ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε αυτή, ο τελάστιος ε, πόρος ε, των εισηγητών θα μπορούσε καλύτερα να, ε, να τύχει διαχείρισης, κάτι το οποίο βέβαια θα σήμαινε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ανατίθενται αυτοί οι πόροι αυτή τη στιγμή και μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο πόρο. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση ε, του χρόνου που περνά από την ε, καταχώρηση, την κατάθεση στη γραμματεία. Ε, κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές το σύστημα δουλεύει όπως θα έπρεπε, αλλά Υπάρχει πολλής χρόνος που περνάει γιατί είναι το προκαταρτικό στάδιο μιας ε, υπόθεσης και αν υπάρχει μια καθυστέρηση στην κατάθεση μιας υπόθεσης, αν υπάρχει μια, ένα διαδικαστικό αίτημα, αν υπάρχει μια υπόθεση η οποία κατατίθεται όχι στη σωστή μορφή και πρέπει να ε, γυρίσει πίσω. Ε, θα με διορθώσει ο συνάδελφος αν κάνω λάθος, γιατί έχει περάσει πολύ χρόνο στο ελεκτικό συνέδριο, όσον αφορά το 63% να σας πω τι ακριβώς σημαίνει αυτό το 63%. Σημαίνει ότι 63, στο 63% των υποθέσεων το, στο δικαστήριο υπήρχε μια καθυστέρηση ε, όχι στο Γενικό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο της Ένωσης. Ε, στο Γενικό Δικαστήριο είναι πιο σύντομη η εκδίκαση των υποθέσεων. για μια διετή υπόθεση θα υπάρχουν δύο ε, διακοπές, ε, Οπότε ίσως να εξηγεί το γεγονός ότι είναι μικρότερη διάρκεια. Δεν υπάρχουν επιπλέον ε, ε, διακοπές. Ξέρουμε ότι οι δικαστικές διακοπές ε, δεν είναι σε κάθε περίπτωση ένα θέμα του κατά πόσο δικαστής είναι εκεί. Μπορεί να μην υπάρχουν επίσημοι, επίσημες διασκέψεις και το λέμε αυτό ε, πήραμε μια απάντηση ας πούμε 14 Αυγούστου, οπότε αυτό σημαίνει ότι κάποιο δούλευε το καλοκαίρι. Δεν ξέρω κατά πόσο ε, μπορεί να αλλάξει αυτό, αλλά με ένα σύστημα που λειτουργεί, σε ένα σύστημα που λειτουργεί με ε, συνεδρίες, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να έχουμε κοινέ διακοπές για όλους τους δικαστές. Ε, το κατά πόσο θα μπορούσε λοιπόν να αλλάξει το σύστημα είναι σχεδόν πολιτικό ζήτημα. Ε, πράγματι μπορεί να υπάρχουν και άλλες βελτιώσεις όπως είπε και η συνάδελφό σας ε, για τους δείκτες τώρα. Κοιτάξτε, το τρέχον σύστημα δεν ε, αξιολογεί τους πόρους που συνοδεύουν μια υπόθεση και πώς έχουν χρησιμοποιηθεί αν ήταν δικηγορικά γραφεία κάθε μισή ώρα θα ήταν κάπου καταγεγραμμένοι. Όμως δεν είναι έτσι το σύστημα. Δεν πρόκειται για δικηγορικό γραφείο. Είναι πολύ διαφορετική η διαδικασία που ακολουθείται. Θα μπορούσαμε όμως να είχε γίνει μια εσωτερική συζήτηση μακροσκελέστερη τι γίνεται με τις μεμονεμένες υποθέσεις και πώς γίνεται η διαχείρισή τους. Αυτό είναι τμήμα της ευρύτερης ε, αναθεώρησής μας. Ρωτήσατε επίσης 84 δικαστές συνολικά, περίπου 400 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Ε, δεν έχω περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με, τους, ε, ε, με, με την αναλογία που με ρωτήσατε. Η κυρία Ντελβό με ρώτησε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό των προσφυγών ω δείκτη, αλλά δεν θα ήταν ο μοναδικό δείκτη. Οι δείκτε δεν είναι το ίδιο πράγμα με του στόχου. Θα μπορούσε να είναι ένα δείκτη, ναι. Ε, δεν ξέρω τώρα έτσι να σας πω πρόχειρα από το μυαλό μου πόσους, ε, πόσες ε, υπάρχουν. Ε, λίγες πάντως είναι, δίκιο έχετε. Θα μπορούσε να υπάρχει λίγο περισσότερη ισορροπία και είναι και ένας δικός μας στόχος αυτό, το δικό μας το συνέδριο, το ελεγκτικό συνέδριο και είμαι σίγουρο ότι και το δικαστήριο θα μπορούσε να το ελέγξει. Όσον αφορά το Brexit, το δικαστήριο πρέπει να το απαντήσει αυτό. Και η ερώτηση του κυρίου λεβγοτόν για τα προδικαστικά αιτήματα και το μέλλον της γαλλικής γλώσσας στο δικαστήριο. Εγώ θέλω να είμαι πολύ σαφής. Ε, στο το, η Daily Mail ε, και διάφορες άλλες τέτοιες εφημερίδες δεν λένε πάντοτε την ε, αλήθεια και με ακρίβεια. Ε, εμείς κάναμε αυτό που μας ζητήθηκε και είπαμε ότι από τη στιγμή που καλύτερη πληροφόρηση είναι, είναι, περισσότερη, είναι περισσότερη πληροφόρηση είναι καλύτερη από τη λιγότερη, έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Ε, υπάρχει επένδυση πολύ μεγάλη στο σύστημα που βασίζεται στη χρήση της γαλλικής γλώσσας ε, όχι ως γλώσσα λειτουργίας του δικαστηρίου αλλά τη γλώσσα των διασκέψεων και λόγω της κλίμακας της επένδυσης αυτής ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα ωφέλη για να υπάρξει αλλαγή. Δεν έχουμε λοιπόν ε, καταλήξει σε κανένα συμπέρασμα. Είναι μια διαδικασία βέβαια που θα ήταν εντελώς διαφορετική. Ευχαριστώ. η κυρία Γκρέσλε. Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ποιο επιθυμεί να ε, αρχίσει. Καλό Εσκομπάρ, εσεί. Ορίστε, κύριε Εσκομπάρ. Καλώ ήλθατε πρώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω γαλλικά για τον κύριο Λεμπροτόν. Θα χαρεί ο κύριος Λεμπροτόν που θα μιλήσω γαλλικά. Αν μου, επιτρέψετε, μου επιτρέπετε, θα ήθελα να τοποθετηθώ σε σχέση με ε, την ε, επισκόπηση, γιατί δεν μπορέσαμε να ε, σχολιάσουμε τις προτάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο αυτό και θα προσπαθήσω να απαντήσω και στις ερωτήσεις που ετέθησαν από ε, τα μέλη και των δύο επιτροπών. Βλέπετε ότι έχω πολύ καλή παρέα σήμερα. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι αυτή η επισκόπηση είναι πραγματικά εξαιρετική στο βαθμό κατά τον οποίο για πρώτη φορά το ελεγκτικό συνέδριο εξέτασε την δικαστική δραστηριότητα των μελών του δικαστηρίου, όχι μόνο την παρακολούθηση δηλαδή της δηλώσεις ε, αξιοπιστίας ε, ε, είναι ακριβώς αυτό που εξετάστηκε είναι πως οι δικαστές ε, διαχειρίζονται τις υποθέσεις, πώς ακολουθούν τους, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν είμαι μόνο η δική μου άποψη, ε, που είμαι ο υπεύθυνο ε, της διαχείρισης των υποθέσεων, αλλά και τα ίδια τα μέλη του, του δικαστηρίου που συμμετείχαν. Εδώ δίπλα μου είναι ο, ο υπεύθυνος του γραφείου ε, και υπάρχει, είναι εδώ μαζί μας και ε, εκπρόσωπος της γραμματείας του δικαστηρίου ε, και εκείνος θα μπορούσε να μας απαντήσει ε, σε κάποιες από τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Ήταν λοιπόν μια ανάλυση αρκετά ιδιαίτερη με γνωρίζουν και οι δύο ε, επιτροπέ. Μιλάω αρκετά ευθέω. Δεν ήταν εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Χρειάστηκε να ε, κάνουμε ε, διάλογο και με τον κύριο Κάρτιφ και με τους συναδέλφους του. Δεν καταλαβαίναμε, για παράδειγμα, πώ το ελεγκτικό συνέδριο είχε επιλέξει τι υποθέσει 600 από τις 2.800 που εκδικάστηκαν σε δύο χρόνια. Για ποιο λόγο η διάρκεια τη της διαδικασίας θεωρήθηκε ουσιαστικός παράγων για την αξιολόγηση της επίδοσης ε, του δικαστηρίου. Εμείς ακούσαμε ποια ήταν η μεθοδολογία, καταλάβαμε ε, τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε το συνέδριο. Υπήρξε όμως ένα πρόβλημα ε, το πρόβλημα είναι ότι στο δικαστήριο υπάρχουν έγγραφα τα οποία καλύπτονται από το απόρριτο των διασκέψεων ή το άρθρο 35 του κανονισμού. Ε, οι διασκέψεις ε, του δικαστηρίου είναι απόρριτες. Αυτό είναι το δίκαιο το πρωτογενέ των συνθήκων, το άρθρο 4, ότι πρέπει να υπάρχει το απόρριτο των διασκέψεων, δηλαδή δεν ε, ε, μπορούμε να δώσουμε ε, κάποια στοιχεία στο ελεγκτικό συνέδριο χωρίς να παραβούμε αυτό το άρθρο. όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία, πρόκειται δηλαδή για στοιχεία για τα οποία δικαστές ή ε, εισαγγελεί παίρνουν μία θέση. Το καταλαβαίνω ότι θα ήταν αυτό πολύ χρήσιμο για το ελεγκτικό συνέδριο για να μπορεί κανείς ε, να εξετάσει το περίπλοκο ε, τη κάθε υπόθεσης, να δει δηλαδή ποια ήταν, ποιο ήταν το πρόβλημα που πραγματεύεται η υπόθεση διαφορά ε, ο κύριος Κάρντι βέβαια με διορθώσει αν κάνω λάθος, ε, υπάρχει ένα σύστημα παράλληλο που δίνει τη δυνατότητα στο ελεκτικό συνέδριο να θέσει απευθείας ερετάσεις, ε, ερωτήσεις ε, στον δικαστή, στο γενικό εισαγγελέα. Μπορούν δηλαδή να μιλήσουν διμερός και νομίζω ότι έδωσε αυτό τη δυνατότητα στο ελεκτικό συνέδριο να έχει τα απαραίτητα στοιχεία, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην ποιότητα της έκθεσης που παρουσιάζει παρουσιάστηκε λοιπόν ήταν ε, πολύ μεγάλη η δουλειά. Νομίζω ότι ε, σωστά διεκπαιρεώθηκε. Ε, τώρα όσον αφορά τώρα τα αποτελέσματα της επισκόπησης, το δικαστήριο ε, επικρότησε τις ε, διαπιστώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Ήμασταν ικανοποιημένοι που είδαμε ότι το ελεγκτικό ε, συνέδριο ανέφερε τις προσπάθειες που κάνουν και τα δύο δικαστήρια να βελτιώσουν το χρόνο επίλυσης των υποθέσεων. Ο κύριος Κάρντιφ φάλωστε, το είπε όσον αφορά τη διάρκεια επίλυσης των υποθέσεων με μείωση αρκετά σημαντική 10 χρόνια περάσαμε από 19,6 σε 14,7 μήνες. Ε, μιλάμε για μέσο όρο διάρκειας και στο Γενικό ε, Δικαστήριο από 28,8 ε, σε 18,7 παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια διεύρυνση το 2004 με νέα ε, δικαστικά ε, συστήματα ε, και αυτό φυσικά ήταν πολύ δύσκολο για μας. Χαίρομαι λοιπόν που έγινε αυτή η παρατήρηση. Ε, δεν μας άρεσε βέβαια που μας είπατε ότι μπορούμε να τα, να, τα, κάνουμε καλύτερα. Μάλλον μας άρεσε που μας είπε ότι μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα, αλλά γιατί πάντοτε μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Ε, ε, γιατί ε, πραγματικά μπορούμε να υποφεληθούμε από αυτήν, ε, αυτό το, το από, την εξωτερική άποψη ε, του ελεγκτικού ε, συνεδρίου. Και κάτι ακόμη, το οποίο εμένα προσωπικά με απασχολεί ε, πάρα πολύ και με αφορά το θέμα της πληροφορικής και της μετάφρασης. Για τη μετάφραση το ελεγκτικό συνέδριο λέει στις υποθέσεις που εξετάσαμε δεν μπορέσαμε να ανοιχνεύσουμε έναν αρνητικό αντίκτυπο σημαντικό στην διάρκεια της διαδικασίας. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει βέβαια, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνο των, ε, των υπηρεσιών ε, ε, μετάφρασης. Λοιπόν, πολύ καλό είναι ότι υπάρχει πολυγλωσία, είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι απαραίτητο, είναι ισότιμη μεταχείριση, είναι δικαίωμα του, του κάθε διαδίκου. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει και η πλευρά της ε, πληροφορικής και μου είπε πολλές φορές ε, ο κύριος Κάρντιφ ε, ότι υπάρχει ένα σύστημα πληροφορικής που έχει κάπως εξελιχθεί αλλά είναι λίγο πρόχειρο γιατί περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία από διάφορες περιόδους. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα πληροφορικής αυτό που έχουμε δρομολογήσει, το γνωρίζετε για να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα από την αρχή της διαδικασίας μέχρι το τέλος και χαιρόμαστε βεβαίως ε, για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μας δοθούν δηλαδή οι πόροι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το εγχείρημα που είναι πολύ σημαντικό. Για τις προτάσεις τώρα τις συγκεκριμένε ε, του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά τη δικαστική εργασία αυτή καθ' αυτή. Και μιλώ υπό τον έλεγχο των συναδέλφων. Λέει το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να έχετε ένα πιο λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, να μην έχετε πολύ γενικό χρονοδιάγραμμα γιατί δεν είναι χρήσιμο, γιατί ανακατεύουμε πιο περίπλοκες υποθέσεις με υποθέσεις που είναι λιγότερο περίπλοκες. Ε, όμως δεχόμαστε μεν αυτή την παρατήρηση, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε από την αρχή αν θα είναι δύσκολη μία υπόθεση ή όχι. Ε, γίνεται, είναι μία ευθεία προσφυγή, ένα προδικαστικό αίτημα και πρέπει να περιμένουμε ήδη το πρώτο ίμιση της διαδικασίας, η έγγραφη να περιμενουμε ηδη το πρωτο ημιση της διαδικασιας η εγγραφη διαδικασια για να μπορούμε να διαβάσουμε ε, τα υπομνήματα των διαδίκων, ε, να δούμε κατά πόσο ε, πρόκειται για προσφυγή, γιατί ακριβώς πρόκειται. Στο τέλος, τουλάχιστον μετά το μέσο της διαδικασίας, θα μπορούμε να ξέρουμε αν είναι δύσκολη ή λιγότερο δύσκολη μια υπόθεση. Ε, ε, κάθε εβδομάδα συνεδριάζουμε, εγώ δεν θα είμαι, σήμερα για παράδειγμα κάθε τρίτη συνεδριάση, που αποφασίζουμε ότι ε, ο σχηματισμός θα είναι πέντε δικαστές, τρεις δικαστές, ε, ένα σχηματισμός μίζωνος σύνθεσης. Ε, είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο να ξέρουμε εκ των προτέρων πόσο δύσκολη και περίπλοκη θα είναι μια υπόθεση, αλλά σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, στο τέλος της έγγραφης διαδικασίας, να μπορούμε να ξέρουμε αν μια υπόθεση θα μπορέσει να επιληθεί πιο γρήγορα, γιατί είναι λιγότερο περίπλοκη και τότε εμείς θα σκεφτούμε ε, τα χρονοδιαγράμματα, τα κάπως πιο ε, προσαρμοσμένα στην υπόθεση. Το κάνουμε ήδη αυτό, το κάνουμε ε, και περάσαμε από τα δύο ε, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ε, σε δέκα από τότε που έγινε η πρόταση του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχει μια πρόταση που σκοπό έχει να υπάρξουν δύο ε, ακόμη χρονοδιαγράμματα ε, για τα ε, προδικαστικά αιτήματα. Μας φαίνεται ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση του ελεγκτικού συνεδρίου. Νομίζω ότι και στο Γενικό Δικαστήριο υπάρχει, και αυτή, και υπάρχει πλέον αυτή η διαδικασία να χρησιμοποιήσουμε ίσως πιο ευέλικτα, πιο αποτελεσματικά τους πόρους διαχείρισης των σπόρων υποθέσεων, το φόρτο εργασίας που μπορεί να εξελίσσεται στα διάφορα τμήματα μεταξύ των διαφόρων δικαστών για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία φάνηκε να είναι προβληματική για κάποιες ε, υποθέσεις γιατί για παράδειγμα απουσιάζει ένα άτομο απρόβλεπτα ε, για παράδειγμα ένα συζητητής ο οποίος αρρώστησε και ε, απουσίαζε για δύο μήνες. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα, έχει αντίκτυπο στη διαδικασία και απρόβλεπτο, είναι κάτι το απρόβλεπτο. Πρόκειται για έναν οργανισμό ε, που ε, δουλεύει ε, συνεχώς και σε, σε, σε, στο 100% είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς κάποιος, να υπο, κάποιον να υποκαταστήσει κάποιον άλλον και είναι δύσκολο να ξέρουμε καν, να ξέρουμε πόσο θα απουσιάσει κάποιο, αλλά το γνωρίζετε αυτό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμβαίνει σε πολλού οργανισμού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή είναι δύσκολο πρόβλημα, ότι δεν μπορούμε να βρούμε μέτρα διαχείριση που να είναι αποτελεσματικά και που να επιτρέπουν να διαχειριστεί κανεί αυτέ τι καταστάσει, να αποφεύγουμε να μπλοκάρει μια υπόθεση για δύο μήνες επειδή ένα συζητητή ε, κολλείεται ή κάποιο δικαστή. Ε, θα το σκεφτούμε, το σκεφτόμαστε ήδη, να ε, ε, μπορέσουμε να το καλύψουμε, να καλύψουμε και πρόταση αυτή. Θα θέλετε να έχετε πιο λεπτομερή στατιστικά, λέει το ελεγκτικό συνέδριο, αξιοποιώντας αυτά τα χρονοδιογράμματα, τα πιο λεπτομερή, τα πιο tailor-made, τα πιο προσαρμοσμένα που μας προτείνεται. Ναι, βεβαίως, στατιστικές ε, που μας δίνουν τη δυνατότητα στα δικαστήρια ε, να οργανώσουν καλύτερα τη δουλειά τους, αλλά και στατιστικές από την άλλη που να μπορούν να ε, ε, δημοσιευθούν για την αποδοτικότητα του δικαστηρίου. Θα έχετε δει εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια στην παρουσίαση των ετησίων εκθέσεων με στατιστικές δικαστικές που είναι όλο και πιο λεπτομερείς και απαντώ εδώ ε, στον κύριο Μαρίνιου Πίντου. Υπάρχουν πολλά στατιστικά στοιχεία τα οποία ήδη υπάρχουν στην ετήσια έκθεση όπως για παράδειγμα τον αριθμό των υποθέσεων ε, που εκδικάστηκαν από ένα συγκεκριμένο σχηματισμό ε, δικαστικό. Νομίζω ότι είναι χρήσιμα και απαραίτητα. Το θέμα τώρα της ευαισθητοποίησης των κρατών μελών ώστε στην ανανέωση των μελών να αποφύγουμε ε, περιπτώσεις ε, να μην ξέρουμε αν κάποιος δικαστής ή γενικός εισαγγελέας που θέλει να παραμείνει, να μην ξέρουμε αν θα μείνει ή αν θα φύγει, γιατί αυτό μπορεί να έχει έναν αντίκτυπο στη διαχείριση των υποθέσεων. Αν θεωρούμε ότι κάποιος θα φύγει, ε, θα σκεφτούμε το τμήμα στο οποίο ανήκει, ότι μπορεί να καθυστερήσει κλπ νομίζω ότι δεν είναι και μυστικό. Ε, και ε, ο πρόεδρος του ε, Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Ένωσης ε, έρχεται σε επαφή με το Συμβούλιο για να τοποθετηθεί το κράτος μέλος σε εύλογο χρονικό διάστημα μερικούς μήνες πριν από το τέλος της θητείας ώστε να μπορούμε να οργανωθούμε και να μην υπάρχει αντίκτυπος στην στη διαδικασία διαχείρισης των υποθέσεων και να την πληρώνουν ε, οι διάδικοι. Το θέμα τώρα των διασκέψεων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, εξηγήσουμε ε, κάτι που το είπε και ο κύριος Κάρντιφ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως πολύγλωσσος οργανισμός και δεν μπορεί να είναι αυτό διαφορετικό. Γιατί είναι δικαίωμα του διάδικου να μπορεί να καταθέσει μία υπόθεση στη γλώσσα του στον κανονισμό της διαδικασίας προβλέπεται αυτό έχει το δικαίωμα να ε, κάνει αγόρευση στη γλώσσα του επακροατηρίου ε, η, η, η η πρωτότυπη γλώσσα πρέπει να είναι η γλώσσα αυτού που καταθέτει ε, την υπόθεση. Αυτό θεωρούμε ότι είναι και θέμα ισότητας μεταχείρισης. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Είμαστε λοιπόν απολύτως πολύγλωσσοι. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι από το 1952, ε, που τότε οι δικαστές αποφάσισαν να ε, μιλούν μεταξύ τους μία γλώσσα, ας κάνουμε μία προσπάθεια να ε, συζητούμε επί τη βάση ενός κειμένου, ας μην χρειάζεται μετάφραση, ας μιλήσουμε σε μία γλώσσα μόνο για μία συγκεκριμένη πρόταση και κατά τη διάρκεια των διασκέψεων δεν υπάρχουν εισηγητές, δεν υπάρχουν διερμηνείς, είναι μόνο οι δικαστές και λένε θα μιλήσουμε μία γλώσσα. Τότε ήταν η γαλλική γλώσσα για διάφορους λόγους, ε, είναι δύσκολο να πάει κανείς πίσω το 1952 να σκεφτεί για ποιο λόγο ήταν τα γαλλικά, ε, όχι τα ολλανδικά, όχι τα ιταλικά, ε, όχι τα γερμανικά. Συγγνώμη, μιλάω πάρα πολύ ώρα να με διακόψετε, αλλά θέλω να σας το εξηγήσω πραγματικά. Ε, διαλέξαμε λοιπόν τα γαλλικά και σύν το χρόνο άρχισαν να έρχονται και άλλοι δικαστές και τέτοιο ζήτημα. Τι θα κάνουμε ε, ε, τώρα. η νομολογία στα γαλλικά είναι απολύτως ακέραιη και δεν θέλουμε τα γαλλικά ε, ήταν η πρωτότυπη γλώσσα και αυτό ήταν κάτι το οποίο οι δικαστές θεωρούσαν πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί όμως να αλλάξει αυτό. Μπορεί οι δικαστές να αποφασίσουν ότι ε, είναι πιο αποτελεσματικό ή είναι πιο βολικό να προσθέσουμε και άλλες γλώσσες που γνωρίζουμε. Οπότε φυσικά ε, στον κανονισμό διαδικασίας μπορούμε να ζητήσουμε μετάφραση ακόμη και για τις γλώσσες για, τις, για τα έγγραφα εργασίας για σα υπενθυμίζω ότι είμαι υπεύθυνο τη μετάφραση, Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να οργανώσουμε ε, τη διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε να τα καταφέρουμε. Θα υπάρχουν βέβαια πλεονεκτήματα, θα υπάρξουν και μειονεκτήματα. Έχουν γίνει συζητήσεις στο παρελθόν, το έχουμε σκεφτεί. Ε, ο πρόεδρος ε, του Γενικού Δικαστηρίου μου είχε ζητήσει διοικητικά στοιχεία και του τα χρωστάω γιατί του τα έχω ε, υποσχεθεί. Κάνω μια, πα, μια παρένθεση για το Brexit. Δεν ξέρουμε φυσικά ποιες ε, θα είναι οι συνέπειες ε, του Brexit στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι ιδιαίτερα πολιτικό και λεπτό το ζήτημα. Ξέρετε ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία τα πιο πολεμικά στην ε, συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν θα υπάρχουν ε, πλέον προδικαστικά ερωτήματα που θα στέλνονται από τους Βρετανούς δικαστές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν υπάρχουν πολλά, θα, θα είναι λιγότερα. Δεν ε, θα υπάρχει ουσιαστικά προσφυγή λόγω παράβαση ε, που ε, θα καταθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι λοιπόν ε, θα έχουμε ουσιαστικά μειωμένες υποθέσεις στα αγγλικά. Τώρα αν θα έχουμε και λιγότερε υποθέσεις στο δικαστήριο, εγώ πιστεύω πως όχι, γιατί πιστεύω ότι θα υπάρξει, μπορεί να υπάρξει μια διαφορά που θα ε, εμφανιστεί και θα σχετίζεται με τον Brexit, δηλαδή πολίτες ε, που θα ζουν στην Ισπανία ή σε κάποια άλλη χώρα και θα απευθυνθούν στον Ισπανό δικαστή για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και αυτό θα καταλήξει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εγώ υποθέτω ότι θα υπάρχουν ε, περισσότερες υποθέσεις αλλά λιγότερες στην αγγλική γλώσσα. Θα εξετάσουμε λοιπόν περισσότερο το στοιχείο αυτό για το θέμα της ενδεχόμενης ε, αλλαγής ε, της γλώσσας των διασκέψεων, όμως ε, το δικαστήριο, αν το επιθυμεί, θα μπορέσει να, επιθυμεί, θα μπορέσει να αποφασίσει σε ποια γλώσσα θα εργαστούν οι δικαστές μεταξύ τους, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και ήδη μίλησα για το σύστημα πληροφορικής, τώρα να πάμε στα άλλα ζητήματα έχω απομακρυνθεί τόσο πολύ που μπορεί να τα ξεχάσω. Λοιπόν, ε, θα φτάσω και στο θέμα της παρουσίας των γυναικών. Ε, ευχαριστώ που μου δώσατε και τα στοιχεία. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουμε πέντε γυναίκες δικαστές ε, και δύο γενικές εισαγγελίες μεταξύ των 39. Ε, τώρα, στην μεταρρύθμιση Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να αυξηθούν οι γυναίκες δικαστές στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης. Κοιτάξτε τώρα, αυτό δεν εξαρτάται ε, μόνο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό δεν εξαρτάται καθόλου από το δικαστήριο. Οι άνθρωποι που προτείνονται, προτείνονται από τα κράτη-μέλη. Εμείς ε, ευχαρίστω να έχουμε όλο ένα και περισσότερε γυναίκε. Ε, αν ισχύσει, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για τα δύο για τον προπολογισμό. Να πάω στον κύριο Μερίνιο Πίντο. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία διαθέσιμα. Μπορούμε να τα προσθέσουμε βέβαια. Έχετε όμω διάφορα στοιχεία στη διάθεσή σα. Θα ήθελα, θα ήθελα αναλυτική πληροφόρηση ο κύριο Μαρίνιο Πίντο. Να επενθυμίσω όμω το εξή. Ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποτελεί το 4% του προπολογισμού των διοικητικών δαπανών της Ένωσης. Είναι το 4%. Αυτός ο αριθμός ε, μένει σταθερός εδώ και χρόνια. Στην πραγματικότητα μάλλον έχει μειωθεί. Το 2010 είμαστε στο 4,13 ενώ τώρα είμαστε στο 4% μετά τη μεταρρύθμιση. Αυτό είναι ο προπολογισμό τη δικαιοσύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήθελα να το πω για να σα δώσω κάποιε αποχράσει. Επίσης, η μεταρρύθμιση που κράτησε τόσα χρόνια από το Μάρτιο του 2011 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ε, το δικαστήριο προσπαθούσε να ανταπεξέλθει ε, σε όλο αυτό τον όγκο εργασίας με μη επαρκή αριθμό δικαστών και ε, για το έτος 2017 είχαμε 3,4 αύξηση του προπολογισμού, για το 2018 θα έχουμε 3,32. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τίμημα για τη δικαιοσύνη, υπάρχει ένα τίμημα, αλλά είναι λογικό το τίμημα σχετικά. Μιλήσαμε για τους εισηγητές. Με συγχωρείτε. Ε, εμείς είχαμε σχεδιάσει μέχρι τις 4 την, πρώτη, ε, την συνεδρίαση αυτή, την κοινή αυτή συνεδρίαση των δύο επιτροπών. Άρα θα πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ και απλώς ε, σας παρακαλώ να το σημειώσετε. Μπορώ να σταματήσω και εδώ, αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε. Απαντάω και στο Σκομπάρ. Ε, φαντάζομαι ότι όσοι υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, αλλά άλλα μέλη έχουν λάβει απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθεσαν. Σεις κυρία Χάουταλα επιθυμείτε να λάβετε το λόγο. Άκουσα ότι είπατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει περισσότερους δικαστές. Από όσο ξέρω, κάναμε μια διοργανική δήλωση. Άρα όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απογοητευθήκαμε ιδιαίτερα όταν είδαμε τις πρώτες, τους πρώτους διορισμούς μετά από αυτό που θεωρώ ότι δεν ήταν ε, έντιμο παιχνίδι. η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας. Αν δεν ήσασταν σημαντικοί δεν θα καθόμασταν εμείς εδώ σήμερα μαζί σας. Και εμείς της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού συζητήσαμε, ας το πω έτσι διπλωματικά, συζητήσαμε επί μια τριετία για το τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω και ορισμένε ερωτήσει, αλλά θα σα τι στείλω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρακαλώ να μου απαντήσετε γραπτώ. Αλλά σα ανακοινώνω από τώρα ότι στα πλαίσια τη ετήσια συζήτηση για την απαλλαγή του προπολογισμού θα επανέλθουμε σε ερωτήσει αυτέ. Δεν μπορούμε να φανταστούμε καν να αντικαταστήσουμε τη γαλλική γλώσσα από την αγγλική και την λέω, τα λέω αυτά στα γαλλικά διότι νομίζω ότι μιλώ καλά γαλλικά. Δεν θα πρέπει να μεταφράζονται τα κείμενα από τα αγγλικά στα γαλλικά και μετά να επαναμεταφράζονται στα αγγλικά. Πρέπει να επιτρέψουμε να λειτουργούν διάφορε γλώσσες, τουλάχιστον αυτέ οι δυο, γιατί δεν εξυπηρετεί η μετάφραση για να ε, δικαιωθεί μόνο αυτή η απόφαση των δικαστών του 1952. Αν και έστω και αν υπάρχει σε ένα κείμενο του 1952. Ε, θα ασχοληθούμε με αυτό και ε, ευχαρίστω θα σας ξανασυναντήσουμε. Πρόεδρος, δυστυχώς και αν το ελεγκτικό συνέδριο δεν θέλει να πει κάτι το απολύτως αναγκαίο για να απαντήσει στα όσα είπε το δικαστήριο. Όχι λοιπόν, καλώς. Θα σας ευχαριστήσω λοιπόν πολύ όλους και τις δύο αντιπροσωπείες από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έλευση σας εδώ και για τις διευκρινήσεις που δώσατε. Ευχαριστώ. The joint meeting is closed. Κλείνει ε, λίγη η κοινή συνεδρίαση.